Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Κοινή συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής προπολογισμών και Ελέγχου του προπολογισμού, Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και όλους. Καλώ ήρθατε κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρία Γεωργίεβα. Και καλημέρα βεβαίως και σε όλους του συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμών. για την Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή αυτός ο προϋπολογισμός που θα είναι στοχευμένο σε αποτελέσματα. Στο άρθρο 83 της συνθήκης υπάρχει από το 2009 νέα διάταξη που ως τώρα δεν έχει υλοποιηθεί. Το άρθρο αυτό απαιτεί λογοδοσία για το τι έχει επιτευχθεί με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και απαιτεί επίσης και εκ των προτέρων καθορισμό της προστιθέμενης αξίας μέσα στα πλαίσια της επικουρικότητας και να αποδεικνύεται γιατί να αναλάβει το ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιο έργο είναι καλύτερο από το να το αναλάβει το εθνικό. Όπως δείχνει και η κατάσταση την οποία ζούμε, αυτό είναι δικαιολογημένο. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πιστεύει ότι η διαδικασία αυτή προσφέρει μια δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει κοινού στόχου και τα βέλτιστα αποτελέσματα κοινού στόχου με τι χώρε μέλη, με το Συμβούλιο των Υπουργών. Ιδίω μάλιστα μέσα σε αυτή την κρίση αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αυτό μα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία. Αντί να συνεχίσουμε λοιπόν business as usual και να αφήσουμε τι χώρε μέλη να πράττουν όσοι έχουν συνηθίσει έω τώρα, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία. Η μέχρι τώρα, ο μέχρι τώρα προσανατολισμό του προπολογισμού μέσω κανονισμών είναι υπερβολικά γενικό ώστε κάθε δαπάνη που ενδεχομένω έχει και εγωιστικό χαρακτήρα αιτιολογείται, δικαιολογείται μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται καλύτερη, καλύτερη κατεύθυνση, καλύτερος προσανατολισμός για να ενισχύσουμε και την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τίθες εκθέσεις πεπραγμένων των γενικών διευθυντών δείχνουν τι έχει επιτευχθεί με τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί ω τώρα. Έχω εδώ αυτό, αυτή τη χοντρή έκθεση που σας δείχνω και με πολύ ενδιαφέροντα παραρτήματα, μάλιστα αν βλέπετε όλο αυτό το έγγραφο, ε, δείχνει τι έχει γίνει με τα χρήματα των διαστατικών ταμείων. Δεν εννοώ ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε λογοδοσία. Υπάρχει λογοδοσία και αυτή είναι η απόδειξη. Γενικέ λοιπόν αιτήσει εκθέσει των γενικών διευθυντών αποκρισταλώνουν καλύτερα το τι έχει επιτευχθεί με τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η δε συνθετική έκθεση του Κολεγίου των Επιτρόπων για όλες αυτές τις εκθέσεις. Όποιος έχει διαβάσει τέτοια έκθεση πραγματικά ξέρει γιατί μιλώ. Τεράστια. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε, να έχουμε το θάρρος να συζητήσουμε και δείκτες αποδοτικότητος και να τους εφαρμόσουμε. Αυτό σημαίνει να δίνεται προσανατολισμός που να ανταποκρίνεται και στις πολιτικές προσδοκίες των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένω με μεγάλη ανυπομονησία την πορεία της σημερινής συζητήσεως, την ε, τοποθέτηση της κυρίας Γεωργίευα. Ευχαριστώ βεβαίως και τις υπηρεσίες μας που κατέστησαν δυνατή την ε, συνάντησή μας αυτή, καθώς και ε, ευχαριστώ και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κυρία Γεωργίευα. Ο κύριος Αρτουή απευθύνω χαιρετισμό στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιφορτισμένη με θέματα των προπολογισμών. Χαιρετίζω και την συναδελφό μου εδώ στα αριστερά μου, πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Χαίρομαι για την παρούσα συνεδρίαση και για τη δημιουργία ενδεχομένω μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τι δημόσιε δαπάνε. Υπάρχει ομάδα υψηλού επίπεδου για του ιδίου πόρου. Θα πρέπει να προσέξουμε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολισμού, που είναι βέβαια μέτριος σε μέγεθος, τελεί υπό τον έλεγχο των χωρών μελών. Θα χρειαστεί λοιπόν ακόμα στενότερη διασύνδεση μεταξύ των δύο επιτροπών μας, ελέγχου του προϋπολογισμού και προϋπολογισμών, μεταξύ ημών λοιπόν και μεταξύ των εθνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών που είναι αρμόδιες για θέματα δημοσιονομικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι η πρώτη συνάντηση που κάνουμε για ζητήματα προπολογισμών μετά τις ε, διακοπές είναι επί των αποτελεσμάτων που προσδοκούμε να επιτύχουμε με τις θυσίες των φορολογουμένων όλοι βλέπουμε πόσο, πόσες κρίσεις μας επηρεάζουν και πόσο σημαντικό είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από κάθε ευρώ το οποίο δαπανούμε. Και αυτό είναι και ο στόχος μας. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε επίγον να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε κάνουμε έχει τις ε, μέγιστες αποδόσεις και την προσθεμένη αξία. Και από την ε, πρώτη στιγμή επικεντρωθήκαμε στις επιδόσεις αυτές ε, στον προπολογισμό, όχι μόνο στις δικές μου υπηρεσίες προπολογισμών, αλλά το κάθε μέλος της ομάδας μας, οποιοδήποτε ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και βεβαίως έχουμε αποφεληθεί στο έπακρον των συζητήσεων με το Κοινοβούλιο και βλέπω εδώ με τα χαράς και τον κύριο Λάζαρο από το ελεκτικό συνέδριο και όπως είπε και ο κύριος Αχτσιβή πρέπει να έρθουμε σε ακόμα στενότερη επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια για να έχουμε μια καλή εικόνα ε, για το πώς θα δομήσουμε αυτό το εγχείρημα και από τους πολίτες μας. Θα επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα. Πρώτον, γιατί ακριβώς έχουμε επικεντρωθεί τόσο πολύ στα αποτελέσματα και τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Δεύτερον, τι πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και ποιες προκλήσεις εντοπίζουμε για το μέλλον. Και τρίτον, κύριοι στόχοι, τι δηλαδή θέλουμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες και χρόνια. Πρώτον, γιατί είναι τόσο σημαντικό. να έχουμε ένα τόσο κυρίαρχο ζήτημα στις συζητήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Κοινοβούλιο και με τα κρατημέλη. Η πρώτη αιτία και πιο σημαντική είναι επειδή αυξάνονται οι ανάγκες ενώ οι πόροι όχι. Σε σχέση με το προηγούμενο ΠΔΠ, οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν συρρυκνωθεί. Και ο μοναδικός τρόπος να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να, να καταφέρουμε να καλύψουμε μεγαλύτερες ανάγκες με λιγότερους πόρους είναι να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε σημαντικά τις επιδόσεις μας. Τον τρόπο δηλαδή που αξιοποιούμε αυτούς τους πόρους. Εδώ βλέπετε και το γράφημα, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Παραπάνω βλέπετε τρεις γραμμές. Έχουμε τις ε, πιστώσεις την κόκκινη γραμμή ε, τις, ε, τις, ε, τις οροφές ε, στις πληρωμών και τα όσα έχουμε κάνει. Για πολύ καιρό παίρναμε πιστώσεις, ενώ ξέρουμε ότι δεν μπορούσαμε να τα ταπανίσουμε όλα αυτά, να απορροφήσουμε όλους αυτούς τους πόρους. Και αυτό έληξε ριζικά με την έναρξη του νέου ΔΠ, είχαμε μια δραματική κρίση πληρωμών και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο γιατί καταφέραμε να βρούμε μία δίωδο και να καταλήξουμε σε έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό. Όμως αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα. Δεύτερον, για πολύ καιρό επικεντρωθήκαμε προβολικά στη συμμόρφωση και στην απορρόφηση, δηλαδή πώς θα δαπανούμε τα χρήματα στο πλαίσιο των κανόνων και δεν είχαμε επικεντρωθεί αρκετά στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Ακριβώς επειδή υπήρχε τέτοια αυθονία που ήταν ε, διαθέσιμη. Τρίτον, κατά τη δέκατη διαπραγματεύσεων για το νέο ΠΔΠ, η συζήτηση αυτή επί των επιδόσεων πήρε σοβαρέ διαστάσει και καταλήξαμε και σε σημαντικέ συμφωνίε. Πρέπει αυτέ τι συμφωνίε να τι υλοποιήσουμε. Τέταρτον, Όπω ανέφεραν και οι δύο πρόεδροι εδώ, υπάρχει ζήτημα και εικόνα, αν θέλετε. Κύρου οι πολίτε μα δεν είναι πεπισμένοι ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που μα δίνουν προ το συμφέρον του. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Κάποιες φορές βλέπουν ότι υπάρχει, βλέπουμε ότι υπάρχει σύγχυση σχετικά με το τι επιτυχάνουμε με τον προλογισμό μας. Και τέλος, είναι σημαντικό όταν υπάρχει εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό γιατί για κάποιους, ειδικά των χαμηλών εισοδημάτων, τους ανέργους, είναι τεράστια ευθύνη για μας να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους προς το συμφέρον αυτών ακριβώς των ανθρώπων. Και εξ ονόματο και των συναδέλφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορώ να σα πω ότι έχουμε πολύ σαφή εικόνα για το πόσο σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στην καλύτερη αξιοποίηση του προπολογισμού μας. Τι ακριβώς επιδιώκουμε λοιπόν με αυτή τη νέα μα προσέγγιση. Εστιάζουμε τις εργασίες μας σε τέσσερις πτυχές. Πρώτον, να είμαστε ξεκάθαρη σχετικά με την προστιθέμενη αξία. Σε ποιους τομείς δαπανούμε, γιατί σε αυτούς τους τομείς είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και όχι τους εθνικούς προπολογισμούς. Τι μπορούμε δηλαδή να προσδώσουμε περαιτέρω από τις δαπάνες σε εθνικό επίπεδο. Μιλήσατε για εγωιστικές δαπάνες, πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εγωιστικές δαπάνες και να αυξήσουμε τις δαπάνες ε, για το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον και το να έχουμε ένα προπολογισμό με προτεραιότητες μας επιτρέπει να σημειώσουμε πρόοδο, κάτι το οποίο έχουμε κάνει, όμως είναι πιο εύκολο να ευθεγραμμίσουμε έναν προπολογισμό με νέες ε, προτεραιότητες και πολύ πιο δύσκολο να τον ευθεγραμμίσουμε με τις περικοπές, να πούμε σε τι δεν θα δαπανίσουμε πλέον. Πρέπει να βρούμε έναν συστηματικό τρόπο να το δομήσουμε. Δεύτερον, πώς γίνονται οι δαπάνες αξιοποιούμε στο έπακρο το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε. Και εδώ πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το έργο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μοχλεύσει ε, περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων μας οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα ευρώ, το κάθε ευρώ, για να προσελκύσουμε και ιδιωτικές δαπάνες. Γιατί πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Πώς απλοποιούμε την εκτέλεση του προπολογισμού. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι το κάθε ευρώ θα αξιοποιηθεί στον ε, προβλεπόμενο σκοπό του και όχι σε διάφορες διαδικασίες που δεν αξιοποιούν σε έπακρον τα χρήματα. Τρίτον, πώς γίνεται η αξιολόγησή μας. Πώς αξιολογούμαστε εμείς οι ίδιοι δηλαδή. Και εδώ θέλουμε πραγματικά να υπάρχει ε, μια αυστηρότατη εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του ελεγκτικού και ρυθμιστικού μας πλαισίου. Γιατί πολλοί λένε αυτή η νέα προσέγγιση που προβάλλεται θέλετε να, ουσιαστικά να αποφύγετε τον έλεγχο προς τη συμμόρφωση. Όχι. Και θα επανέλθω. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα επιπλέον στοιχείο στις μετρήσεις μας, ούτως ώστε να ε, καταγράφουμε καλύτερο τρόπο τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Και αυτό βεβαίως είναι συναφές με οποιαδήποτε αλληλεπίδρασή μας με το Κοινοβούλιο και με τις επιτροπές ε, που ασχολούνται με τα ζητήματα των προπολογισμών. Με την ετήσια διαδικασία προπολογισμών και για, τις, ε, για την ενδιάμεση αναθεώρηση και με τα μετατοπή ΔΕΛΤΑΠΗ. Και για την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ιδίους πόρους, να πω ότι εκτός και αν καταφέρουμε ξεκάθαρα να αποδείξουμε τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού προπολογισμού, πολύ δύσκολα θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση για τους ιδίους πόρους. Και ο Υπουργός Σόιμπλε, πάντα θυμάμαι ότι λέει, αν θέλετε να αλλάξουμε τον κύκλο εσόδων του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει πραγματικά να αποδείξετε τα ωφέλη από, τις πλευράς, από πλευράς δαπανών. Δηλαδή, αν το αποδείξετε αυτό, θα καταφέρουμε να αυξήσουμε και τους ίδιους πόρους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ήδη κάνουμε πολύ σημαντική δουλειά στον επόμενο κλάδο, το πώς ακριβώς κοινοποιούμε και επικοινωνούμε αυτές μας τις προσπάθειες. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Ό,τι κάνουμε υπάρχει κάπου ως πληροφορία. Όμως, κάποιες φορές είναι θέμα οργάνωσης είναι τόσο δύσκολο να το βρει κανείς. Ιδίω για τους πολίτες μας. Είναι δύσκολο να κατανοήσουν τι ακριβώς κάνουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ενοποίησης πολλαπλών βάσεων δεδομένων που δείχνουν τα αποτελέσματα ε, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, αλλά ελπιστούμε ότι θα μας οδηγήσει σε μια καλύτερη πλατφόρμα για να μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία. Τι έχουμε κάνει, πόσε θέσει απασχόληση έχουμε δημιουργήσει, πόσο έχουμε βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον, πόσο έχουμε βοηθήσει του γεωργού μα, πώ έχουμε βοηθήσει του εθνικού προπολογισμού να είναι πιο διαφανεί και καθαρότεροι, πόσο έχουμε συμβάλει στην καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου κλίματο, όλα αυτά τα στοιχεία. Προχωρώ στο επόμενο. Τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Τι πρόοδο υπάρχει γιατί παρότι ως δομημένο τμήμα του έργου μας αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε βασιστεί σε προηγούμενες προσπάθειες, τις οποίες και συνεχίζουμε. Έχουμε ένα σύστημα μέτρησης και κοινοποίησης ε, των παρελθοντικών εργασιών. Αυτό έχει ενσωματωθεί και στα νέο ΠΔΠ. Βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωση, αλλά ήδη εντάσσεται στι διαπραγματεύσει σε αυτό το τμήμα. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Στο νέο ΠΔΠ πραγματικά υπάρχει σημαντική εστίαση στα αποτελέσματα και επιδόσει. Εντό των παραμέτρων ε, των προπολογισμών, όπω γνωρίζετε και εσεί κύριε Αχτσουή στην επιτροπή σα, είχαμε μεταφέρει κονδύλια προ ε, την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Με πολύ μικρό περιθώριο ε, όπου καθορίζεται το 80% του προπολογισμού, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να στραφούμε και προς άλλες και νέε προτεραιότητες. Στο νέο ΠΔΠ εργαζόμαστε με πολύ καλύτερο τρόπο για πολλαπλούς ε, στόχους. Το 1 ευρώ με ένα σμπάρο δύο τριγώνια θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τέλο πάντων δεν είναι πολύ ε, οικολογική παρατήρηση. Με το 1 ευρώ επιτυχάνουμε περισσότερο από έναν στόχο στο κλίμα για παράδειγμα, μπορούμε να επενδύσουμε στην ενεργειακή απόδοση, ω εκ τούτου να βελτιώσουμε τι οικονομικέ επιδόσει, να αυξήσουμε την απασχόληση, δημιουργία θέσεων απασχόληση ε, για μικρέ επιχειρήσει που α πούμε κατασκευάζουν υποδομέ. Ταυτόχρονα επιτυχάνουμε και του ε, οικολογικού περιβαλλοντικού μα ε, στόχου για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Με ένα πολύ απλό παράδειγμα, δηλαδή βλέπετε ότι καταφέρουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα κρίση στο γάλα, κρίση προσφυγική. Βλέπουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους γεωργούς αλλά και τους πρόσφυγες και όσους χρειάζονται επιγόντως τροφή. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε περαιτέρω και να καλλιεργήσουμε ως φιλοσοφία. Γι' αυτό και είμαι και επίτροπος αρμόδια για το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί αυτά πρέπει να γίνουν οριζοντίως. Μα απασχολεί ιδιαίτερα η υψηλή μόχλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ήδη αναφέρθηκα στο ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά και στο κόσμο και σε άλλα μέσα. Υπάρχει διασύνθεση με την οικονομική απόδοση, δηλαδή για τα προγράμματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια με έναν τρόπο ώστε να υποστηρίζονται οι ευρύτεροι στόχοι για αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα και μεταρρυθμίσεις. Επίσης, ανάλογα με τις επιδόσεις, έχει κάποιος πρόσβαση σε επιπλέον κονδύλια. Αν κάποιος θα πηγαίνει καλά, θα πάρει και προσθέρα χρήματα δηλαδή. Αλλιώς αυτά τα χρήματα θα πάνε σε προγράμματα με καλύτερες επιδόσεις. Και βεβαίως, μας απασχολεί ιδιαίτερως και το, τα απλοποιημένα σύστημα, συστήματα παράδοσης. Τώρα, για τη μείωση του σφάλματος, του ποσοστού σφαλμάτων. Είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε πάντα να περιορίσουμε το ποσοστό σφάλματος σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά μας. Και εν συντομία να αναφέρω και δύο παραδείγματα. για τα όσα εμείς εντοπίζουμε ως ε, δείκτες επιδόσεων και εδώ υπάρχει σημαντική βελτίωση έχουμε αυξήσει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην έρευνα. Είναι κρίσιμη σημασία στοιχεία για την οικονομία μας, αλλά και για να σταματήσει αυτή η λεγόμενη διαρροή εγκεφάλων προς τις ΗΠΑ, που είναι πολύ έντονη τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μας βοηθήσουν ε, σε αυτό το σκοπό. Μετά, το χαμηλό κόστος ε, σύστασης επιχείρησης. Αυτό είναι ο στόχο μα. Ιδίω ό,τι αφορά τι startups, θέλουμε να του επιτρέψουμε να κινούνται πιο γρήγορα, χωρί ε, υψηλό κόστο και διοικητικό άκθο. Νέε θέσει απασχόληση για του ερευνητέ. Το βραβείο Νόμπελ του 2014 ιατρικής. Σαφή σύνδεση μεταξύ ε, επενδύσεων και υψηλότερων επιδόσεων. Απασχολησιμότητα στο Erasmus Plus. Τι σημαίνει και μετρούμε δηλαδή, τι σημαίνει το να κινείται κάποιο από τον ακαδημαϊκό χώρο στην αγορά εργασία και είναι σαφή τα ωφέλη. Σε διεθνέ επίπεδο, καταπολέμηση του έμπολα, ανθρωπιστική βοήθεια σε Συρία και Ουκρανία, χρηματοδότηση περιβαλλοντική. Αυτά είναι παραδείγματα όπου μπορούμε να μετρήσουμε με μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματά μας και τις επιδόσεις μας. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Βεβαίως ε, τώρα βρισκόμαστε στις αρχές ή μάλλον στα μέσα του δρόμου. Ελπίζω να μας βοηθήσει και μια συζήτηση που θα κάνουμε στη συνέχεια. Δεν είναι εύκολο να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Πρώτον, δείκτες. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τους δείκτες, τι είναι ρεαλιστικό και τι όχι. Τι κόστος είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε για την τελειοποίηση των δικτών. Σε ποιο σημείο θα πούμε εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ. Είναι αρκετά καλοί οι δείκτες μας. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να αντλήσουμε από αθρηστικά στοιχεία συμπεράσματα τα οποία να, είναι, να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται και ε, σε μεμονωμένες ε, δραστηριότητες. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η διασύνδεση αν θέλουμε να είμαστε και φτηνοί και αποτελεσματικοί, πώς γίνεται αυτό, γιατί έχουμε και θετικές και αρνητικές εμπειρίες. Τι μπορούμε να κάνουμε, τόσο αυτή η διαχείριση με βάση τις επιδόσεις, να κινηθεί ταχύτερα σε ό,τι αφορά τα ε, προγράμματα και την ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Ουσιαστικά θέλουμε να βελτιώσουμε τη δικασία λήψη αποφάσεων ε, και την ε, συλλογή των στοιχείων που μας οδηγεί σε αυτή την λήψη αποφάσεων. Και βεβαίως εσείς μας βοηθάτε μόνο και μόνο που μας ενημερώνετε για τις ε, δράσεις σας και που μας ελέγχετε. Γι' αυτό είναι πολύ καλό για το Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερως, γιατί ξέρω ότι υπάρχει προβληματισμός. Το να στραφούμε προς τις επιδόσεις σημαίνει ότι αποφεύγουμε τον, ε, την εστίαση ως προς τη συμμόρφωση. Και αυτό δεν ισχύει. Για το ποσοστό σφάλματος στο πλαίσιο των ε, επιδόσεων. Έστω, όπως ισχύει και σήμερα, γιατί εμείς θέλουμε το ποσοστό σφάλματος να λάβει ένα δίκτυο ο οποίος ε, τηρείται. Αλλά ας πούμε ότι και πάλι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό αυτό. Έχουμε πολλές ενέργειες για περαιτέρω απλούστευση, επιπλέον ελέγχους ε, που επικεντρώνονται στην ε, σχέση κόστους-οφέλους ε, και περισσότερες μεταρρυθμίσεις και σε επίπεδο κρατών μελών. Επομένω, επανασχεδιάζουμε προγράμματα και ενδεχομένως να λαμβάνουμε και δημοσιονομικές αποφάσεις βάσει επιδόσεων. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πούμε ότι δεν πρέπει να διαθέτουμε τόσους ε, πόρους εκεί, γιατί δεν υπάρχουν ε, τα απαραίτητα αποτελέσματα. Τώρα, πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα. Έχουμε δύο σημαντικές χρονικές στιγμές για μάθο μέλλον. Πρώτον, έχουμε τη συνδιάσκεψη για τη νέα προσέγγιση αυτή στις 22 Σεπτεμβρίου επικεντρωνόμαστε στα, ε, στις επιδόσεις και είναι πολύ σημαντική αυτή η συνδιάσκεψη. Θέλουμε να αποτελέσει μια ευκαιρία αλλαγής. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε πρόβλημα. Ήταν η μοναδική ημερομηνία που μπορούσαμε να κλείσουμε μεγάλη αίθουσα. Έπρεπε λοιπόν να την κλείσουμε, αλλά σίγουρα του χρόνου αυτό δεν πρόκειται να συμβεί θα βρούμε τρόπο να ενημερώσουμε στο έπακρον όποιον ενδιαφέρεται. Βεβαίω λογικό είναι, φέτο ε, θα επικεντρωθούμε στι επιδόσεις ε, στον δημόσιο τομέα και τα όσα ξέρουμε από την πράξη. Νέε επιδόσει, ε, προοπτικές, στόχοι για τον προπολογισμό και τι επιδόσει και θέλουμε να μιλήσουμε και για τι επιδόσει στον τομέα του κλίματο. Γιατί πλησιάζει και η διάσκεψη του, των Παρισίων. Θα είναι υψηλού επίπεδου η διάσκεψη. Περιμένουμε και υπουργού και ευρωβουλευτέ, το ελεγκτικό συνέδριο. Όλοι οι αρμόδιοι επίτροποι θα παρίστανται και ο Ζαν Κλοντ γιουγκερ θα κάνει την κύρια ομιλία. Και μάλιστα τώρα ακριβώ ε, κάνουμε μια συζήτηση και με ρωτάει τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε. Μετά τη συνδιάσκεψη θα έχουμε ένα πιο λεπτομερές ε, σχέδιο δράσης. Η, δεύτερη σημαντική διάθρωση είναι η ομάδα για, την, ε, για τον προπολογισμό που είναι βασισμένο σε αποτελέσματα. Θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στην ουσία με μια σύνθεση της ομάδας αυτής που να είναι ευρεία αλλά και διαχειρίσιμη. Και αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε. Και ένα κοινό όραμα για την εργασία στον τομέα αυτό. Ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να συνθέσουμε τη διαθεσμική ομάδα. Θα απευθύνω λοιπόν έκκληση προς όλες και όλους να εξευρεθούν οι αναγκαίες συμβιβασμοί, ώστε η εργασία αυτή να μπορέσει να αρχίσει και στα σοβαρά. Έχουμε ομάδα εργασίας των επιτρόπων για την performance, για την απόδοση και όντως εντυπωσιάζομαι από τη δέσμευση και από την ποιότητα εργασίας των επιτρόπων. Με συγχωρείτε, μακρυγόρισα ίσως λίγο, αλλά μου φάνηκε ότι θα είναι σημαντικό να σας εξηγήσω την διάθρωση των όσων προσπαθούμε να επιτύχουμε, καθώς και τον τρόπο σκέψης μας. Η Συμπρόεδρος κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε για την πρώτη αυτή ματιά που μας επιτρέψατε να ρίξουμε στο συνεχιζόμενο έργο σας και εγώ εκφράζω τη λύπη μου που δεν θα είμαστε παρούσες στις 22. Θα βρούμε τρόπο πάντως να επικοινωνούμε και να ενημερωνόμεθα. Τώρα, για, την, για το θέμα των error rates θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, κύριο Λαζάρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ελεγκτικό συνέδριο καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε ένα performance-based budgeting. Είναι η σωστή κατεύθυνση, διότι όπως έχουμε πει σε ορισμένες από τις εκθέσεις μας, πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο στην απόδοση και ταυτόχρονα βέβαια με την βελτίωση της συμμόρφωσης. Με το έργο μας εμείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεχίζουμε να συμβάλλουμε προς την επίτευξη, επίτευξη, προς την επίτευξη μάλλον καλύτερων αποτελεσμάτων μέσα στα πλαίσια πάντα και της συμμόρφωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν και ρητή ευλογία των εργασιών μας από το ελεγκτικό συνέδριο. Θα δώσω το λόγο τώρα στις πολιτικές ομάδες. Η γραμματεία έχει χωρίσει τις πολιτικές ομάδες αρχίζοντας με τον συντονιστή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού μετά ε, αναλόγως ε, οι συντονιστές ώστε να έχετε περίπου μια ιδέα πότε θα έρθει η σειρά σας και μετά από τους συντονιστές θα λάβουν, ε, θα λάβουν τα μέλη το λόγο, οι ευρωβουλευτές δηλαδή, για ένα λεπτό. Χωσέ Μανουέλ Φερνάνδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένα ορόσημο για το μέλλον και κάθε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι κάθε ευρώ του προϋπολογισμού που βγαίνει από την τσέπη του φορολογούμενου θα πρέπει να επιστρέφεται, να έχει ανταπόδοση και να ελέγχεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού για να ξέρουμε πού χρησιμοποιήθηκε το κάθε ευρώ. Γι' αυτό θα ήθελα να σας συγχαρώ και να υποβάλω και ορισμένες ερωτήσεις. Θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι η επίδοση είναι η εκτέλεση ο δείκτης εφαρμογής, ο δείκτης εκτέλεσης. Εμείς ορίζουμε ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με βάση τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και για να έχουμε μια καλή επίδοση, καλές επιδόσεις, θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, ε, την απασχόληση δηλαδή το στόχο καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, του στόχου στην παιδεία, στην καταπολέμηση της φτώχειας. Εμείς ορίζουμε στόχους και μετά λέμε ότι για αυτούς τους στόχους έχουμε μία ποσοστιαία αναλογία του προϋπολογισμού για την πλήρωση αυτών των στόχων. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει σωστή επίδοση, δηλαδή κατά πόσο έχουμε φτάσει σε αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ένα πολύ καλό πι στο μέλλον. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ε, ζητώ συγγνώμη. Έχετε ένα λεπτό ο καθένας, μόνο μία πρόταση, μία. Μία πρόταση μόνο. Αυτό, αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική για την αναθεώρηση του ΠΔΠ. Τη στιγμή που έχουμε προγράμματα για την εκτέλεση και έχουμε και ένα πρόβλημα με τις ε, πληρωμές. Δεν μπορούν να υπάρχουν καλές επιδόσεις εάν δεν υπάρχουν οι κατα... κατάλληλες επιστώσεις. Ορίζοντας 2020 ε, δεν έχει σωστή εκτέλεση γιατί δεν έχει τους κατάλληλους πόρους. Είμαι πολύ κακό παράδειγμα. Κακό παράδειγμα ήσασταν για την τήρηση του χρόνου. Ο κ. Σάβαμα τώρα, της Επιτροπής Ελέγχου. Ε, μια στιγμή να βρω και το σωστό μικρόφωνο. Ήδη μου κόστησε αυτό λίγα δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ αγαπητοί συμπρόεδροι. Εσείς ευχαριστώ και εσάς κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Να μην χάσω χρόνο λέγοντας ευγενικά λόγια καλύτερα να ρίξω το βάρος μου σε αυτή την στάση που ε, έδειξε και η ίδια η κυρία Γεωργίευα που λέει ανασκουμποθείτε και δουλέψτε. Και βλέπω τη στάση της αυτή από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι το εξής. Πρέπει να αρχίσουμε τη δουλειά, να εξετάσουμε τους δείκτες. Να μην τους κάνουμε και υπερβολικά περίπλοκους και να ρίξουμε τη ματιά μας στα δεδομένα των χωρών μελών και στο ποσοστό σφάλματος. Να δούμε πού δαπανώνται τα χρήματα. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα δύσκολο και περίπλοκο. Όλο αυτό το σύστημα με τις χιλιάδες ε, διάβλους που έχουμε γύρω μας το κάνει δύσκολο αυτό, αλλά ε, να φανούμε γενναίοι, να ε, προσπαθήσουμε να βρούμε το δρόμο μας μέσα από αυτή τη ζούγκλα. Να δούμε ποια είναι η πραγματική απόδοση, πού πάνε τα χρήματα και τι επιτυγχάνουν. Ούτε κι εσείς ήσασταν καλό παράδειγμα για την τηρήση του χρόνου, λέει η πρόεδρος Γκρέσλετ. Τώρα ένα λεπτό η Ινιές Αιάλα Σέντερ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επίτροπο για αυτή την πρωτοβουλία που μας ε, βοηθά, όπως είπε και ο κύριος Φερνάντες, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να τηρήσουμε. Θα πρέπει όμως να βελτιώσουμε την, ε, το ποσοστό των δίκτυ εφαρμοσιμότητας και εφαρμογής. Δεν σε συμφωνώ γιατί όπως έχει λεχθεί θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η ομάδα ανθρωπίνων πόρων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη νύχτα των ε, κρυστάλλων όπου έχουμε ένα πολύ λυπηρό ε, και ξέρουμε ότι ο κύριος ε, Σόιμπλε και το παρελθόν του ορίζουν αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να δώσουμε εξηγήσει στους ε, πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε πληροφόρηση, επικοινωνία και απλούστευση, γιατί εδώ έχουμε μεγάλα ελλείμματα. Και θα πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα με τους πολίτες. Θα πρέπει κάθε ευρώ των εθνικών προϋπολογισμών να δαπανάτε καλά. Αυτό ισχύει και για τον κοινωτικό προϋπολογισμό. Σχεδόν καλό παράδειγμα. Ρουμπιάλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα μπω στην ουσία. Συμφωνώ με την ανάγνωση του ζητήματος που κάνετε. Δηλαδή θα πρέπει να βελτιώσουμε τον ε, ευρωπαϊκό προπολισμό με δύο κόκκινες γραμμές. Μιλάμε για μια σωστή εξισορρόπηση και χρήση των ε, διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι πολλά μέτρα οικονομικά δεν είναι βιώσιμα, αλλά κοινωνικά είναι αναγκαία. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, τύχουν υποστήριξης. Καταρχήν υπάρχουν οι πολιτικές ε, όχι σκοπιμότητες αλλά ανάγκες και φοβάμαι γιατί ορισμένα προγράμματα δεν λειτουργούν αλλά εάν υπάρχει πολιτική βούληση θα βελτιώσουμε το πρόγραμμα για να επιτύχουμε το στόχο. Γι' αυτό οι πολιτικές προτεραιότητες έχουν άμεση σημασία γιατί πιστεύω ότι υπάρχει άμεση αναγκαιότητα εφαρμογής των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Πολύ καλό παράδειγμα ήσασταν εσείς για το ECR. Εσείς, Ρίτσαρτ, ναι. Ναι, εγώ, εγώ, εγώ είμαι. Δεν προβλεπόμουν, αλλά εγώ θα λάβω το λόγο. Καταρχήν, Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Μιλήσατε για την ουσία ναι, αυτό είναι ένα πολύ ογκώδες ζήτημα και θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίσουμε τις προτεραιότητες σε σχέση κόστους ωφελίας και πώς θα χειριστούμε αυτό το οικοδόμημα του προϋπολογισμού το οποίο καταραίει. Δεύτερον, ως προς τη διαδικασία έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στα σφάλματα, στο περιθώριο σφάλματος και θα πρέπει να ε, φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης και να ε, επανορίσουμε το πρόγραμμα για την αναγνωρισιμότητα των σφαλμάτων. Θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τη μέτρηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων με την άρση προσκομμάτων έτσι ώστε οι Ε να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα. Αν θέλουμε μηδενικό ποσοστό σφάλματος τότε τα προσκόμματα θα είναι πολύ υψηλά. Και τρίτον, το οικοδόμημα δεν θα είναι πλήρες μέχρι ότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει υψηλότερη εποπτεία. Έχουμε εκλεγεί άμεσα και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις επιδόσεις ακόμα. Και αυτό είναι ο, ο κρίκος ο οποίος λείπει στο όλο οικοδόμημα. Και εσείς υπερβήκατε το χρόνο. Τόιρε από τις φιλελευθέρους δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος από τους ε, φιλελευθέρους που θα το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι κατά πόσο θέλουμε ένα προϋπολογισμό που να βασίζεται στις επιδόσεις, διότι το, το εγχείρημα είναι πολιτικό και όχι τεχνικό. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, χρησιμοποιείται ε, για να λιπάνει ένα μηχανισμό ώστε να υπάρχει πραγματικά πραγματική εκτέλεση. Αν δούμε τις αιτήσιες εκθέσεις από το ελεγκτικό, ε, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι καταστροφική ως προς τις επιδόσεις. Ε, δεν λαμβάνεται υπόψη ο κοινοτικός προϋπολογισμός και αυτό οφείλεται στα κράτη λέμε για περιορισμένα χρήματα, αλλά αν δούμε τις, ε, την ε, μεταποιητική βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, έχουμε 5,6 δις ε, διαφοροποίηση της οικονομίας, 5 δις χωρίς καμία προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Μιλάμε για 10 δις που είναι 20% του ΑΕΠ του Λουξεμβούργου. Άρα το ζήτημα είναι κατά πόσο θέλουμε έναν προϋπολογισμό που να βασίζεται στις επιδόσεις. Εγώ τον το επιθυμώ, γι' αυτό και είχα υποβάλει τροπολογία για τη διαδικασία απαλλαγής πέρσι και είπαμε ότι ως Κοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε μία ομάδα υψηλού επίπεδου για τις επιδόσεις. Λυπάμαι, αλλά είμαστε γραφειοκράτες, τίποτα άλλο. Λυπάμαι που είμαι όμως, αλλά θα πρέπει να ε, το θέσουμε πολιτικά το θέμα. Θέλουμε ένα προϋπολογισμό που να βασίζεται στις επιδόσεις πραγματικά. Φιλελεύθεροι τώρα, εσείς από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Και εσάς βεβαίως ε, κυρία Αντιπρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη νέα σας αυτή πρωτοβουλία για την διαμόρφωση του προϋπολογισμού βασισμένου σε αποτελέσματα, ένα από τα προβλήματα ήταν ότι μέχρι τώρα ο προϋπολογισμός στόχευε κυρίως την απορρόφηση των κονδυλίων, χωρίς να έχουμε πραγματική δυνατότητα και λογοδοσίας και ελέγχου των αποτελεσμάτων. Άρα βρίσκω αξιέπαινη την πρωτοβουλία σας. Υπάρχουν και ορισμένοι λόγοι που καθιστούν πάρα πολύ σημαντικούς τους δείκτες για την μέτρηση της αποδοτικότητας. Χωρίς δείκτες δεν μπορούμε να μετρήσουμε την αποτυχία ή έστω τα επιτυχημένα αποτελέσματα. Και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων καθίσταται ανεπεριεχομένου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Ένωσης απέναντι στα μάτια του κοινού να υπάρξει ο έλεγχος αυτός. Γι' αυτό και λέω και πάλι ότι η πρωτοβουλία σας είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Τώρα σχετικά με την διαθεσμική ομάδα εργασίας που προτίθεστε να ε, δημιουργήσετε. Τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Η εντολή και οι στόχοι της ομάδας αυτής έχουν καθοριστεί ορθά. Ωστόσο αυτό που με ανησυχεί είναι περισσότερο η συχνότητα των συνεδριάσεων της ομάδας αυτής θα παρουσιάσει τα πρώτα της αποτελέσματα σε τέσσερα χρόνια. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα επανεξετάσετε. Τώρα έρχεται η Ενωτική Αριστερά. Δεν γνωρίζω το όνομά σας, με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει. Δεν πρόκειται για επιχείρηση λογοδοσίας. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι αυτοί που χρησιμοποιούν τα χρήματα. Μιλούμε για δημόσιες δαπάνες και πώς θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τους λαούς της Ευρώπης, καθώς επίσης για διαχείριση των σπάνιων πόρων, που μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν στοχεύσουμε στους στόχους, στους ε, στόχους για την απασχόληση, αξιοπρεπή απασχόληση, αντιμετώπιση της φτώχειας, παιδεία και σε ό,τι αφορά τους πολλαπλούς στόχους. Να ληφθεί υπόψη είναι και το ζήτημα της ισότητας των φίλων και να μην μείνει μόνο στα λόγια. Ούτε από τους στόχους αυτούς τελικά να υποφεληθούν μόνο οι τράπεζες τα δεδομένα πρέπει να μετρώνται καλύτερα. Δεν έχουμε τις διάφορες λεπτομέρειες, τις αποχρώσεις και πώς μπορούν να μετρώνται αυτές. Υπάρχουν λοιπόν ανάμεσα στα δεδομένα σημαντικές αποκλήσεις. Πρέπει να γίνουν συγκρίσιμα για να ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά μας εν τέλει. Ε, ευχαριστώ λέει η πρόεδρος Κρέσλε. Δεν βλέπω τον κύριο Ντε Ιόγκ. Υπάρχει κανείς ε, που να τον, αντιπροσωπεί, να τον ε, συγγνώμη. Τώρα εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν αρκεί βέβαια η χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού, δεν αρκεί η απορροφησή τους, πρέπει να μπορεί να ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο απορροφώνται. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε δείκτες. Οι δείκτες αυτές πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι και να μην αμφισβητούνται το να μιλούμε για αποδοτικότητα των δαπανών κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ γενικά. Χρειάζονται δείκτες και υποδείκτες που να δείχνουν ακριβώς τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει αποδοτικότητα. Με την έννοια αυτή μπορούμε να υποβάλουμε και τους δείκτες αυτές σε ένα διαρκές monitoring. Και βεβαίως πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα τι γίνεται εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι που μετρώνται με τους δείκτες. Το θέμα λοιπόν τότε τίθεται της απαλλαγής. Ευχαριστώ πραγματικά υπόδειγμα τη ρίσος του χρόνου. Η πράσινη τώρα κύριο Στάραντ. Ρωτήσατε, ρώτησε κάποιος πριν, θέλουμε performance based budgeting. Εγώ ασφαλώς και θέλω. Τώρα, κοιτάξτε, πριν από δύο χρόνια έγινε μια συνάντηση μεταξύ μου και ενός ανώνυμου γενικού διευθυντή, τον οποίον ρώτησα εάν στην μακρά του σταδιοδρομία στα θεσμικά όργανα είχε περάσει και καμιά επιτυχία. Και μου είπε, αφού σκέφτηκε καλά, ναι, δύο φορές δεν μπόρεσα να ταπανίσω όλα μου τα κονδύλια. Τι να σας πω, καλή τύχη στην προσπάθειά σας να αλλάξετε την αποτροπή αυτή. Η FTD. Ζάνη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ εντάχει. Δέχομαι την πρωτοβουλία αυτή. Είναι ευπρόσδεκτη γιατί θα πρέπει να έχουμε δείκτες επιδόσεων, συγκεκριμένους δείκτες που είναι απολύτως αναγκαίοι και για τη δική μας Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και γενικότερα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα είναι ένα μέσο για τα κράτη-μέλη για να έχουν μία σαφέστερη ιδέα ως προς την εφαρμογή των πολιτικών τους, διότι πολύ συχνά έχω την εντύπωση ότι στο Συμβούλιο ε, δεν υπάρχουν ε, σαφή ιδέα για το που οδεύουν. Τώρα ε, εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί μέχρι τώρα δεν βασιστήκαμε στις επιδόσεις. Μέχρι τώρα δεν κάναμε τίποτα για αυτό το θέμα. Ίσως ε, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ελπίζω να υπάρχει η βούληση, αυτό το βλέπουμε εδώ και θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα θεσμικά όργανα. Εντάχει, ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο που είναι εδώ και μας παρουσίασε το πρόγραμμά της. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε την προστιθέμενη αξία το, της χρήσης των πόρων και των ταμείων. Αυτό το βλέπουμε και από το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί και ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ είπε ότι σήμερα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μόνο ένα προϋπολογισμό που είναι η συσσόρευση όλων των εθνικών προϋπολογισμών. Θα πρέπει να άρουμε την πελατιοκρατία που υπάρχει μέχρι τώρα. Θα πρέπει οι επιδόσεις να συμβαδίζουν με τη διαφάνεια. Είναι κάτι που μας απασχολεί εμάς τους πολίτες. Vielen Dank. Die ENF von Ali. Ευχαριστώ. Από την TNF. Καλά. Κύριε Επίτροπος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητος αυτός ο διάλογος. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πολιτικά θέματα, αλλά και θεσμικά, το οποία θέλουμε να λάβουμε υπόψη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα σχόλια και ερωτήματα που θέσατε και χρήζουν απάντηση. Ξεκινώ από το ζήτημα της ε, κατανομής. Πράγματι έχουμε την Ευρώπη 2020. Είναι κοινή στόχη για όλους, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέσω εθνικών προγραμμάτων, προς τα οποία συνεισφέρει και ο ευρωπαϊκός προπολογισμός. Και εκεί υπηρετεί το θέμα της κατανομής, γιατί είναι μόνο 1% του ε, ΑΕΠ ο υπερπολογισμός, Επομένω, το θέμα είναι πώ θα μετρήσουμε ακριβώ τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από το ευρωπαϊκό προπολογισμό που είναι τόσο μικρό σε σχέση με του ε, εθνικού και πώ μετρούμε και τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει σε σχέση με του δικού μα στόχου. Ο προπολογισμό μα βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων ε, και αντιστοιχεί στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γιούνκερ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μας και επίκαιρο θέμα, το οποίο έχουμε συζητήσει και με το Ευρωπαϊκό Ολυμπικό Συνέδριο. Γιατί αν κάνουμε το λάθος να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε πώς αυτή η πολύ μικρή συμβολή του προπολογισμού οδηγεί ή όχι στην ε, μείωση της ε, ανεργίας, για παράδειγμα, σε, με αριθμητικά στοιχεία, αυτό είναι λάθος. Αλλά αν πούμε, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, έχουμε διάμεσους δείκτες να μετρήσουμε την επιτυχία, τότε αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου. Παρεπτόντως, γιατί κάνουμε αυτή τη διάσκεψη και ξεκινούμε με τις πρακτικές και την πρακτική μας εμπειρία. Γιατί ήδη υπάρχει τέτοια εμπειρία για το τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνεται. Τι είναι σφάλμα αν θέλετε. Όμως, κύριε Φερνάντες, έχετε δίκιο. Πρέπει να πούμε αυτές είναι προτεραιότητες, αυτός είναι ο προπολογισμό συμβάλλει προς αυτές τις προτεραιότητες και πώς μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη συμβολή. Μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές αυτό το ε, πλαίσιο ενημέρωση, κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και, και το καθεξής. Γιατί αν εμείς επιτυχάνουμε αποτελέσματα αλλά δεν το μαθαίνει ποτέ κανένας ή τα ερμηνεύει εσφαλμένα, τότε δεν ακολουθούμε τη σωστή προσέγγιση. Και είναι σημαντικό να λέμε τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό και τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει σύγκληση ή όχι. Ή απόκληση. Και τι ακριβώς ε, κερδίζουμε από όλο αυτό. Για τις κόκκινες γραμμές είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα ότι τελικά πρωταρχικός μας στόχος είναι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες δυνάμεις στον κόσμο είναι αποτελεσματική και το έχουμε καταφέρει γιατί είμαστε και κοινωνικά υπεύθυνη οντότητα μέχρι τώρα. Έχουμε αυτή τη φήμη και αυτή τη φήμη οφείλουμε να την διατηρήσουμε. Προφανώς, αν πούμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και αυτό δεν μεταφράζεται σε θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας, αυξάνονται τα κέρδη, αλλά αυτό δεν έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως λοιπόν. Το μόνο που ήθελα να πω και αυτό κάπου αναφέρθηκε στη συζήτηση. Α, ναι, στη δική σας ε, παρέμβαση. Κάποιες φορές ενδεχομένως να χρειαστεί να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα έχει πολύ υψηλό ποσοστό σφάλματος. Δεν παρέχει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά ωφέλη. Ίσως ε, να είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά δεν πρέπει εμείς να το χρηματοδοτήσουμε, γιατί δεν είναι καλά τα αποτελέσματα. Ίσως πρέπει να πάει σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Και γι' αυτό απαιτείται και μια δόση ειλικρίνειας για το πώς εμείς ε, αξιολογούμε τη συμβολή μας και την προσταθεμένη αξία μας. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χθες ήμουν στη Βουλγαρία, την πατρίδα μου, για τα εγγένεια μιας ε, μεγάλης μονάδας διαχείρισης ε, απορριμμάτων, μία από τις ε, μεγαλύτερες στον κόσμο. Εκεί υπήρχε και ένα ζήτημα για κατά πόσο αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό ή από τον εθνικό προπολογισμό. Γιατί να χρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ένα τέτοιο πρόγραμμα στη Σόφια, που είναι μια αρκετά πλούσια πόλη, να θέλετε, σχέση με άλλες πόλεις στη Βουλγαρία. Και η απάντηση είναι απλή. Γιατί η συμβολή του ευρωπαϊκού προπολογισμού οδηγεί σε αλματώδη ανάπτυξη. Αντί η να ε, μείνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, το πώς ε, θα φτιάξουμε τη χωματερή, τι θα γίνει κτλ, πέρασε σε άλλο επίπεδο. Καλή ποιότητα, καλή οικονομική επίδοση, οι δείκτες. Αυτό δεν θα γινόταν χωρίς τη δική μας εμβολή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, συγγνώμη που επιμένω. Ο Πρωθυπουργό τη Βουλγαρίας μου είπε πριν από 5-10 χρόνια θα πήγαινα στη Βιέννη για να δω μια τέτοια μονάδα. Και τώρα οι Αυστριακοί θα έρχονται στη Βουλγαρία να δουν τη δική μα μονάδα γιατί είναι καλύτερη. Κατά σύμπτωση και ο επικεφαλής, η επικεφαλής ε, της μου είναι Αυστριακή και του είπα, της είπα ορίστε να δεις εσύ. Αλλά αυτό εντάξει το είπα στη ευόμενη. Όμως αυτή η προσταθήμενη αξία της αλματόδους ε, μετακίνησης είναι κάτι που πρέπει να γνωρίσουμε ως ε, θετικό επίτευγμα ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Πρέπει να πούμε τι συμβαίνει με ευρωπαϊκά κονδύλα που δεν θα μπορούσε να γίνει με εθνικά και αν γίνεται κάτι καλύτερα με τα ευρωπαϊκά από ό,τι θα γινόταν με τα εθνικά κονδύλια, θα πρέπει να υπάρχει τόπο να το αναφέρουμε και αυτό. Τώρα, αν χρειαζόμαστε πραγματικά διαμόρφωση του προπολογισμού με βάση τι επιδόσει. Και πολλοί απάντησαν ήδη σε αυτό το ερώτημα, πράγματι χρειάζεται. Να αντιστρέψω μάλιστα το σχόλιο αυτό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση value for money και μέτρηση των επιδόσεών μας. Ιδάλλως, οι πολίτες μας δεν θα μας στηρίξουν και αν δεν μας στηρίξουν ένας μεγάλος παράγοντας ε, επιτυχίας της Ένωσής μας θα επανομευθεί. Θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί τρελό σήμερα. Δεν αποκλείω ακόμα και να ζητήσουμε μεγαλύτερο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιους τομείς ανταγωνιστικού πλονεκτήματο ή ε, ισχύω. Σκεφτείτε τι κάνουμε ακριβώ τώρα με την προσφυγική κρίση. Αλλά πρέπει να το αποδείξουμε αυτό με στοιχεία ότι είμαστε οι πιο αποτελεσματικοί για την αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Θα είναι απαραίτητο, αλλά δεν θα συμβεί αν δεν το αποδείξουμε. Για να σας απαντήσω λοιπόν, και βλέπετε και τα φώτα που αναβοσβήνουν, δείχνουν ότι έχει έρθει η ώρα της αλήθειας. Είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ενδιαφέρον ήταν το ζήτημα της ε, απόδοση ευθυνών τη λογοδοσία, ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίω θα πρέπει να το διαρευνήσουμε. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και όλο το θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουμε επιτροπέ ε, του Κοινοβουλίου, υπάρχει λογοδοσία και στο δικό μα τον προπολογισμό, τον εσωτερικό. Όλα αυτά πώ ακριβώ ε, σε λειτουργούν. Και ίσω ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργούμε καλύτερα. Αλλά δεν θέλω να ξεφύγω από το σχολείο σας. Το έχουμε συζητήσει. Εμείς θεωρούμε ότι όσο περισσότερη λογοδοσία υπάρχει, τόσο το καλύτερο γιατί έτσι βλέπουν και οι πολίτες ότι παίρνουμε στα σοβαρά ε, τα συμφέροντά τους και λέμε και εμείς τι έχουμε κάνει. Είναι σαφές το μήνυμά σας ότι είναι η αξιοποίηση των πόρων και είναι και ένας ε, τρόπος ε, να μειώσουμε και τις απώλειες να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε την ανισότητα στις κοινωνίες μα, Τα άκουσα όλα αυτά και τα σημείωσα τα μηνύματά σα. Βεβαίω ε, και ο δρόμος και ο τρόπο που θα ε, δομήσουμε ακριβώ ε, αυτού του δείκτε είναι σημαντικό θέμα. Ήδη έχουμε κάνει πολλά και θα επανέλθουμε και στο μέλλον. Πάντα βεβαίω εγώ κάνω την εξή έκκληση. Πάντα Πρέπει να λέμε όχι τι καλό θα ήταν να γίνει, αλλά τι πρέπει να γίνει για να γίνει σωστά η δουλειά. Και τέλος, μην νομίζετε ότι θα υπάρχουν αποτελέσματα για τους πάντες. Γιατί εκεί θα χαθούμε. Εμείς το αντίθετο θέλουμε να κάνουμε. Να λέμε λίγες βασικές προτεραιότητες και μετά να δούμε, να μετρήσουμε πώς ε, λειτουργήσε ο προπολογισμός θα ήθελα να συνεχίσουμε το διάλογο αυτόν και για διαιτερότητες, πιο συγκεκριμένους τομείς για παράδειγμα, να πούμε τι έχει αλλάξει χάρη αυτό, σε αυτή τη νέα προσέγγιση. Και κάτι τελευταίο, χρησιμοποίησα αυτό το residual rate στην ομιλία μου. Ξέρω ότι το Ελληνικό Συνέδριο έχει δική του εντολή γι' αυτό. Είναι σημαντικό να έχουμε μία αξιόπιστη μέτρηση του ποσοστού αυτού σφάλματο και αυτό γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάληψη δράση, η οποία είναι πάντα σε συνάρτηση με το ποσοστό σφάλματος. Αν λάβουμε, αναλάβουμε δράση θα μειωθεί το ποσοστό σφάλματος. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να αναλαμβάνει ο κόσμος δράση και γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το ποσοστό σφάλματος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλο το πλαίσιο του πώς επικεντρωνόμαστε στις επιδόσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Η πρόκληση βεβαίω τώρα είναι να είμαι εξίσου αποτελεσματικό με την κυρία Γκράσλε. Σημείωσα ότι οκτώ μέλη μα έχουν ζητήσει το λόγο. Υπενθυμίζω ότι θα πρέπει ε, να περιουστείτε στο ένα λεπτό. Έκαστος. Η κυρία Μουτή. Thank you. Uh, I'll do my best. Ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Χαιρετίζω ιδιαίτερως ε, αυτή τη στόχευση στην αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία. Ότι δηλαδή αξιοποιούμε στο έπακρο αυτά τα χρήματα και τα κονδύλια για να προσφέρουμε κάτι παραπάνω στην οικονομία. Αλλά και τα όσα είπατε ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται στο έπατον και συμφωνώ απολύτως, χαίρομαι που αναφερθήκατε στην έρευνα και στο βραβείο Νόμπελ. Έχω και εγώ κάποιες και συμμερίζουμε κάποιες ανησυχίες ότι κινούμαστε προ τη μόχλευση και ότι η μόχλευση θεωρείται προσωπική αξία και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξεχάσουμε και τη σημασία της άμεσης χρηματοδότησης. Μιλήσατε Ε, ε, μάλλον εγώ διερωτώ αν έχετε ασχοληθεί εγκαρσίως με το θέμα της ε, ισότητας των φύλων. Και τέλος, για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την προσέγγιση που αναφέρατε για τον προπολογισμό σε ένα μέσο και όχι σε ένα αυτοσκοπό. Και αν δούμε για παράδειγμα ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πώ καταλαβαίνουμε αν δεν λειτουργεί καλά επειδή μήπω δεν έχει υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυστοφόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ ότι τα πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματο, άρα είμαστε υπέρ τη ε, να υπάρχουν και δείχτε απόδοση και επιδόσεω για να μπορούμε να μετρούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των κονδυλίων. Σίγουρα ένα προπολογισμό των 150 δισεκατομμυρίων για κάποιο είναι πολύ μικρό, είναι το 1% των προπολογισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για πολλού άλλου είναι μεγάλο γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο από πολλού προπολογισμού των χωρών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που θέλουμε να ξέρουμε από αυτά τα 150 δισεκατομμύρια θα φτάνουν τελικά εκεί στο σκοπό στον οποίο απευθύνονται. Και αυτό που έχει αξία και σημασία και δεν το λαμβάνουμε υπόψη είναι η γραφειοκρατία. Πόσο κόστο πληρώνουμε για γραφειοκρατία και πόσα αφαιρούνται από τον προπολογισμό. Απίφθηνα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξίζει τον κόπο να την αναφέρω ποια ήταν η απάντηση στι 8 Σεπτεμβρίου, όπου μου αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με βάση το τυποποιημένο μοντέλο κόστου η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι διοικητικέ επιβαρύνσει που απορρέουν από τι νομοθεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για 13 επιλεγμένου τομεί προτεραιότητας ανέρχονται σε 124 δισεκατομμύρια ετησίω. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε και στο ζήτημα τη γραφειοκρατίας εάν θέλουμε πραγματικά αυτοί οι δείχτε να έχουν και αυτή η απόδοση και επίδοση. Merci. Madame Thomas. Η κυρία Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πίτροπε για την παρουσία σας. Όπως είπατε οι επιδόσεις είναι πολύ σημαντικές. Ε, μέσα σε ένα λεπτό δεν μπορώ να σας δώσω τη γνώμη μου. Θα κάνω τρία σχόλια. Εάν οι επιδόσεις σημαίνουν μείωση της γραφειοκρατίας που προπετείται από την Κομισιόν και τη μείωση του κόστους διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων, τότε τάσσομαι υπέρ γιατί δυστυχώς στη δική μου εκλογική περιφέρεια πολλοί οργανισμοί και ενώσεις μου λένε και ιδιαίτερα άνεργοι ότι δεν ζητάμε ε, επιδότηση από το ΕΚΤ διότι μας στοιχίζει πολύ περισσότερο να κάνουμε την αίτηση. Εάν επίσης θέλουμε να επαληθεύσουμε ότι οι πόροι πάνε ε, εκεί που πρέπει και όχι στις μεγαλύτερες διαρθρώσεις που έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τους φακέλους, αυτό θα ήταν πολύ καλό. Τέλος, ερώτηση. Εάν υπάρχει ε, κακή εκτέλεση ή αποδοτικότητα, ας πούμε στην ενεργεία των νέων, εάν το μέσο εγγύηση για τους νέους δεν λειτουργεί, τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε ε, την τάξη πραγμάτων, εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Ολμπριχτ. Ευχαριστώ. Ορισμένα σχόλια και μόνο. Κύριε Επίτροπε, υπάρχει ένας κίνδυνος. Εάν μιλάμε για προϋπολογισμό βάση επιδόσεων, ε, καλύπτουμε όλο, όλα τα πεδία. Τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, αποδοτικότητα και ε, όλα τα σχετικά. Διαφορετικά χάνουμε το χρόνο μας δεν μιλάμε μόνο για τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, γιατί δεν είμαστε ε, παράρτημα του ελεγκτικού. Μιλάμε για τη διαδικασία διαχείρισης του προϋπολογισμού. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τους ε, δείκτες. Οι δείκτες δεν πρέπει να έρθουν μετά τον προϋπολογισμό, αλλά με τον προϋπολογισμό. Άρα, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να αλλάξουμε τη συλλογιστική μας. Βον. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το τελευταίο σημείο του Γιάννα, όλοι καλωσορίζουμε αυτή την μέτρηση της απόδοσης ή αποδοτικότητας και το ελεγκτικό. Είπε ότι δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι αριθμοί, αλλά η μέτρηση των επιδόσεων. Είχατε συζητήσεις με το ελεγκτικό συνέδριο για να ξέρουμε ότι ε, έχουμε την ίδια θεώρηση. Ως προς την ομάδα υψηλού επίπεδου, είπατε ότι στην Επιτροπή θα θέλατε να συνεργαστείτε με αυτή την Επιτροπή και υπάρχει καθυστέρηση από το Κοινοβούλιο. Έτσι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Μπορείτε να μου πείτε αν αληθεύει αυτό. Thank you. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, εποπτεύει τον ε, προϋπολογισμό και αυτό είναι πολύ σκόπιμο γιατί ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν δαπανηθεί καλά τα χρήματα. Εάν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση ότι για κάθε project θα πρέπει να υπάρχουν εκ των προτέρων κρατήρια, τότε ε, αυτό θα ήταν ε, πολύ καλό. Δηλαδή θα ξέρουμε ότι είναι ένας ευφυής τρόπος μέτρησης εκ των αποτελεσμάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο το ελεγκτικό να μας δώσει ε, αριθμητικά στοιχεία για δείκτες επιτυχίας ε, ή αποτυχίας. Εάν είχαμε ένα τέτοιο αριθμητικό στοιχείο από το ελεγκτικό, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς και να ξέρουμε πού γίνεται κακή χρήση ή δαπάνη των χρημάτων. Τον Άνω. Αυτή η συζήτηση τον αυτη άκρος ενδιαφέρουσα Θέλουμε να μειώσουμε τους δείκτες ε, σφάλματος, να υπάρχουν καλύτερες επιδόσεις και αποδοτικότητα. Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά ποια Ευρώπη θέλουμε. Θέλουμε μία Ευρώπη των καθολικών αξιών που είπε και η κυρία Γεωργίεβα. Θέλουμε να υπάρχει ποιότητα ζωής για τους πολίτες μας. Θέλουμε να υπάρχει κοινωνική πρόοδος θέλουμε αυτή την αναγνώριση. Αυτά είναι τα ζητήματα ουσίας. Και βεβαίως και τα λογιστικά είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι το ουσιώδες. Τι επιδόσεις θέλουμε για τους πολίτες μας. 48 δευτερόλεπτα, μπράβο. Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν, δεν επιδέχεται περαιτέρω γραφειοκρατία. Δεν ξέρουμε πόσα χρήματα προβλέπονται για του, για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Δεν ξέρουμε πόσα χρήματα παίρνει το κάθε ε, ταμείο. Μιλάμε για την ανεργία των νέων, αλλά δεν ξέρουμε πόσα χρήματα ε, προβλέπονται για αυτή την περίπτωση. Αυτό το χάσμα θα πρέπει να το καλύψουμε. Υπάρχει άμεση σχέση και αιτιώδη συνάφεια θα μπορούσα να πω μεταξύ γραφειοκρατίας και εκτέλεσης των ε, προγραμμάτων. Αυτό το βλέπουμε και με τα στοιχεία που έχουμε για την Ιταλία το 2006. Η Ιταλία είχε χιλιάδες project τα οποία δεν μπορούσε να ελέγξει. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε με μικρά project θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Χρειαζόμαστε δείκτες απόδοσης, για παράδειγμα για την ΕΕΒ έχουμε τα δεδομένα των πρέσβεων σε σχέση με την χρήση των πόρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις εκθέσεις για τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολισμού θα μπορούσαμε να συνδράμουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω το εγχείρημά σας, κυρία Αντιπρόεδρε, και θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις κι εγώ οι επιδόσεις από την πλευρά των κρατών μελών θα πρέπει να οδηγήσουν στο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, τα καλύτερα δυνατά. Ο ρόλος μας δεν είναι εύκολος. Βλέπουμε πώς έχει θεσμική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που έχει σημασία είναι να χρηματοδοτήσουμε και μικρά projects. Αλλά όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε, όσο πιο μικρά είναι τα project, τόσο υπάρχει περισσότερο κίνδυνος ε, απάτης. Γι' αυτό τι κάνουμε. Επιβαρύνουμε τη γραφειοκρατία και δημιουργούμε μια πολύ κακή εικόνα για την Ευρώπη. Γιατί ότι μιλάμε για 4-5 ε, ευρώ και έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε με μια Ευρώπη ε, υπερβολικής γραφειοκρατίας. Δηλαδή δημιουργούμε ένα χαρτομάνι άνευ προηγουμένου. Ας πούμε για την περίπτωση των ε, προσφύγων. Χρειαζόμαστε περισσότερες πιστώσεις, αλλά πώς θα έχει η αποδοτικότητα τη στιγμή που τα κράτη-μέλη έχουν το προνόμιο της υποδοχής των προσφύγων και των μεταναστών. Άρα μπορούμε να ζητήσουμε από τους αρχηγούς κρατών να ανταποκριθούν. Και στη συνέχεια θα ήθελα να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς εξελίσσονται οι δείκτες επιδόσεων. Υπάρχει αυτή η μανία των δικτών. Τα αποτελέσματα δεν είναι τα καλύτερα δυνατά ως προς τη μείωση των δημοσίων δαπανών και του δημοσίου ελλείμματος. Ας μειώσουμε αυτό το χαρτομάνι, αυτό το reporting, ε, από το οποίο δεν βγάζουμε τίποτα αλλά φυσικά το εγχείρημα έχει μεγάλη σημασία και μπορούμε να επιταχύνουμε και το χρονοδιάγραμμα. Γιατί αν θα πρέπει να ελέγξουμε τις δημόσιες δαπάνες, δεν θα πρέπει να έχουμε ένα πενταετές ε, πρόγραμμα. Θα πρέπει τους επόμενους μήνες να έχουμε τις ε, πρώτες προτάσεις. Η κυρία Γεωργίεβα για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για τα δικά σας σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω για το ρόλο των δικτών. Αρκετοί ομιλητές στο δεύτερο γύρο ανέφεραν κάποιες επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τη χρήση των δικτών. Και δικαίως. Εάν περάσουμε σε μια μηχανιστική προσέγγιση, όπου απλώς ε, συλλέγουμε αριθμητικά στοιχεία για δεδομένα και μένουμε μόνο σε αυτά, δεν θα λειτουργήσει καλά το σύστημά μας, για δύο λόγους. Πρώτον, οι δείκτες έχουν περιορισμούς. Δείχνουν μόνο εν μέρη. Τι κάνουμε για να πετύχουμε ένα στόχο. και σε ιδεατέ συνθήκε, Δηλαδή, α πούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα απασχόληση και βεβαίω το μετρούμε με τον αριθμό των θέσεων απασχόληση που δημιουργήθηκαν. Όμω, αν δημιουργούνται χαμηλή ποιότητα, χαμηλά αμοιβόμενε θέσει εργασία ή ε, θέσει που στο τέλο του προγράμματο θα εξαφανιστούν, τι ακριβώ σημαίνει το αριθμητικό στοιχείο, πώ ε, θα μετρήσουμε και την ποιότητα του έργου μα, είναι πολύ δύσκολο και νομίζω ότι ο κύριο ε, αυτή πολύ σωστά τα ανέφερε. Είναι και πολιτιστική δηλαδή η αλλαγή, η αλλαγή νοοτροπίας. Να σκεφτόμαστε τα αποτελέσματα, όχι μόνο το πώς θα διώξουμε τα χρήματα. Ακούσαμε και το παράδειγμα του Γενικού Διευθυντή που είπε ότι απέτυχα δύο φορές, δεν μπορούσα να ταπανίσω τα κονδύλια που μου αναλογούσαν. Ίσως ήταν και πολύ καλό βέβαια, γιατί σημαίνει ότι έκανε πολύ καλή αξιοποίηση των χρημάτων του. Δεν το ξέρουμε όμως, γιατί δεν έχουμε αυτή την οτροπία να σκεφτόμαστε τα αποτελέσματα. Η ευθυγράμμιση όμως με τις προτεραιότητες είναι κάτι που αποδεδειγμένα λειτουργεί. Και υπάρχουν και άλλες δυσκολίες, δηλαδή το πώς οι αριθμητικοί δείκτες με τους περιορισμούς τους μπορούν να μας βοηθήσουν. Η απάντηση είναι σε αυτό που είπατε νομίζω. Πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την προσέγγιση, να ε, μεριμνούμε για τα χρήματα των φορολογουμένων μας. Σε συνδυασμό και με τους δείκτες που χρησιμοποιούμε και η συνάδελφός μου η Νάντια Κολβίνο είπε ότι δεν είναι ένα μηχανιστικό σύστημα. Η αφοσίωση για τις επιδόσεις είναι αυτή που μας οδηγεί. Βεβαίως θα υπάρξουν ευκαιρίες να προσδιορίσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα όταν έχουμε και προσανατολισμό με βάση τις επιδόσεις με τους περιορισμούς που προκύπτουν και από τα μειονεκτήματα των δικτών αλλά θα είναι πολύ καλύτερο από το να μην ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Πάντα δίνω αυτό το παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε έναν δρόμο με μηδενικό ποσοστό σφάλματος αλλά δεν οδηγεί πουθενά. Είναι λοιπόν 100% καλή χρήση ε, των πόρων ή 100% σπατάλη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σπατάλη. Επομένω, το να φύγουμε από αυτή την προσέγγιση είναι μόνο εάν πραγματικά η νοοτροπία μας μας επιτρέπει να επικεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα. Άκουσα το μήνυμα να μην είναι το, η μοναδική μέτρηση, η μόχλευση. Βεβαίως και όχι. Όμως, το ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια μας πιο αποτελεσματικά για να αυξήσουμε την ιδιωτική επένδυση στην οικονομία μας σε μια χρονική στιγμή που οι ιδιωτικοί επενδυτέ φοβούνται τον κίνδυνο, είναι ένας καλός στόχος. Ένας από τους πολλούς βέβαια, όχι μοναδικό. Τώρα, αν κάνουμε προπολογισμό με βάση τη διάσταση του φύλου, ναι. Ε, λίγο περισσότερο δυστυχώ ε, στην εξωτερική διάσταση, στα ανθρωπιστικά, στα αναπτυξιακά, περισσότερο υπάρχει εκεί, αλλά είναι και περισσότερο το εντάσσουμε και στην εκτέλεση του δικού μας υπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προσπαθούμε να δούμε ε, εάν ε, βελτιώνουν τη θέση της γυναίκας ε, στο χώρο εργασίας, οι συνθήκες πώς είναι. Το εξετάζουμε, αλλά βεβαίως δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μας. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ε, θέμα της συμμόρφωσης που ανέφερε ο κ. Όλμπριχ και βεβαίως ε, των δικτών. Και στην αρχική μου παρουσίαση ανέφερα πώς ακριβώς ε, θα αξιολογήσουμε τη σχεση κοστος κόστους-οφέλους. Και δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει βεβαίως. Συνεργαζόμαστε με το Ελληνικό Συνέδριο από αυτού ε, ήρθαν σε επαφή μαζί τους και με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι θέλουν να συμμετάσχουν και στην ε, διαθεσμική ομάδα. Βεβαίω βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία. Ελεγκτικό συνέδριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο κοινό. Θα ήταν πολύ αρνητικό εάν καταλήξουν σε μια μεθοδολογία το ελεγκτικό συνέδριο και σε άλλη μεθοδολογία η Κομισιόν. Πρέπει με κάποιον τρόπο να συγκεράσουμε τι καλύτερε εμπειρίε, του καλύτερου εμπειρογνώμονε. Βεβαίω υπάρχει ανεξαρτησία από πλευρά του. Εμεί έχουμε τι υποχρεώσει μα. Αλλά πρέπει να το οδηγήσουμε προ μια κοινή κατεύθυνση το θέμα. Και επ' αυτού εκτιμώ ιδιαίτερω αυτή την ευκαιρία που έχουμε να συνεργαστούμε. Δεν λέω ότι θα επιβραδύνουμε την ομάδα του επίπεδου εξαιτία αυτή τη νέα ε, Εξέλιξη, Έχει το χρονοδιάγραμμά του η ομάδα αυτή και θα συνεχίσει τι εργασίε τη. Και εδώ και ο Μάριο Μάντι συμφωνεί ότι η ομάδα του επίπεδου έχει μεγάλε πιθανότητε επιτυχία να αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο ε, παράγονται έσοδα για τον προπολογισμό, εάν ταυτόχρονα αυξήσουμε και την εμπιστοσύνη στην ε, επιτυχή αξιοποίηση των πόρων μας. Αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν είναι αλληλένδετα, αλλά δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα. Και έτσι θα κλείσω με αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Ανεβάζουμε τα μανίκια και ξεκινάμε δουλειά. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Καταλάβαμε ότι για να επιταχυνθούν οι ρυθμοί των εργασιών της ομάδος εργασίας για τους ιδίους πόρους θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Αν προχωρήσουμε γρήγορα μπορεί και ο Μόντι λοιπόν να αποφασίσει να επιταχύνει. Μάλιστα, αυτό υπόσχεται πολλά. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι η αποτελεσματικότητα της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών χρειάζεται μια διαρκή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και, ελέγχου, και, ε, και Επιτροπής Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Γεωργίευα. Ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών τη Επιτροπή προπολογισμών σε 5 λεπτά 10 και 40 λέει ο πρόεδρο, που είναι 9 λεπτά.